Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την, ε, της της πρώτης ομάδας εργασίας, προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών, Ευρώπη των αξιών και των δικαιωμάτων. Μόλις με ενημέρωσαν ότι ο εισηγητής μας, ο κύριος ε, Λόπες Αγγιλάρ, έρχεται, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών. Θα ήθελα καταρχάς να χαιρετήσω τον Πιέρ Λικηγέ που είναι συμπρόεδρος. Το πρόφερα καλά, πολύ καλά. Θα προεδρεύσουμε με κάθε αλληλεγγύη σήμερα το απόγευμα σε αυτήν την ομάδα εργασίας. Κάθε ένας από τους δυο μας θα κάνει μια σύντομη εισαγωγή και θα δώσουμε τις απόψεις μας ε, για το θέμα της ομάδας εργασίας και συνεχεία θα δώσω το λόγο στους ε, ομιλητές, σε όποιον τον θέλει και στο τέλος ο εισηγητής, ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ, θα καταλήξει κάποια συμπεράσματα και θα συνοψίσει τις εργασίες της ομάδας εργασίας. Αυτή είναι η μερίσια διάταξη της, των εργασιών μας, αν συμφωνείτε. Κύριε Λεκυγέ, θέλετε να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ, Σοφή. Θα ήθελα να σας πω ότι μου φαίνεται πολύ σημαντική αυτή η ομάδα εργασίας. Πολύ σημαντική γιατί όταν μιλάμε για την Ευρώπη, συχνά αναφέρουμε το νόμισμα, την οικονομία, την καταπολέμηση της λαθομετανάστευσης κτλ. κτλ. Αλλά δεν μιλάμε για τις αξίες. Και νομίζω ότι η Ευρώπη οικοδομείται πάνω σε αξίες. Και έτσι οικοδομήθηκε μέχρι στιγμής. Το κοινοτικό κεκτημένο αυτό είναι ένας πραγματικά τεχνοκρατικός όρος. Είναι πάντως το γεγονός ότι 27 χώρες συμφώνησαν μέσω της νομοθεσίας τους για να προωθήσουν κάποιες κοινέ αξίες. Νομίζω ότι για να μιλήσουμε στους πολίτες, το γεγονός ότι έχουμε κοινέ αξίες, το γεγονός ότι υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι υπάρχει το, η Χάρτα των Θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχει νομική και δεσμευτική αξία. Τουλάχιστον σε 24 από τις 27 ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά έχουν απήχηση στο μυαλό και στην καρδιά των Ευρωπαίων πολιτών. Και νομίζω ότι πέρα από την οικοδόμηση του χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας επί του οποίου εργαζόμαστε με τρόπο πολύ θετικό μέσω της Στοκχόλμης, μέσω και πέρα από τις ε, εξουσίες που θα πάρουμε και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτόν τον τομέα, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για δικαιώματα και για αξίες στους πολίτες. Θα πρέπει να ανυψώσουμε τη συζήτηση και να απευθυνθούμε στο συνέστημα των ανθρώπων. Υπάρχουν δικαιώματα και αξίες που κατέχει η Ευρώπη και που οι άλλοι ήπειροι δεν έχουν όταν κάνω ομιλίε μπροστά σε νέου Ευρωπαίου πολίτε, του λέω ότι η Ευρώπη έχει τι δικέ της αξίε. Και μία από τι προποθέσει, παραδείγματο χάρη για να μπει κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η κατάργηση τη θανατική ποινή. Όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε αποφάσισαν και όλε όσε θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισαν να αποποιηθούν ε, αυτή τη ποινή, κάτι που δεν υπάρχει σε πολυάριθμες άλλες χώρες και είναι ένα θέμα επί του οποίου θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση για να πείσουμε και άλλους να σταματήσουν να εφαρμόζουν αυτή την ποινή. Μαζί με τη Σοφή λοιπόν θα συμπροεδρεύσουμε σε αυτή την σύνοδο. τη δίνω ξανά το λόγο ούτω ώστε να ξεκινήσει έτσι η συζήτηση. Έχουμε ήδη τρία αιτήματα για συζήτηση ο κύριος Κάλης, μετά τον κύριο Λόπες Αγγιλάρ. Σας ευχαριστώ. Τώρα, ε, η δική μου αρχική παρέμβαση. Πιστεύω και ελπίζω ότι έχουμε αρκετή τροφή για συζήτηση, αρκετά θέματα για συζήτηση, γιατί αν όλοι συμφωνείτε, αν όλοι συμφωνούσατε μάλλον, δεν έχει νόημα συζήτηση, δεν θα μπορούσαμε σπίτι. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη των δικαιωμάτων και των αξιών, Νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν θέματα για συζήτηση γύρω από αυτό το πλαίσιο, μέσα από αυτό το πλαίσιο. Α είμαι λίγο προκλητική, έτσι για να δρομολογήσω λίγο τη συζήτηση. Άκουσα κάποιε από τι παρεμβάσει στην ε, προηγούμενη σύνοδο τη Ολομέλεια και άκουσα μερικού να λένε ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να λέει τίποτα για τι αξίε και για τα θεμελιώδη δικαιώματα, γιατί είναι εθνικό θέμα. Και η Ευρώπη απλώ θα πρέπει να ασχολείται με τεχνικά θέματα, με τα θέματα της εσωτερικής αγοράς κτλ. Ε, θεμελιωδώ, ε, ε διαφωνώ κάθετα με αυτό το θέμα. Γιατί αν έχει κάποιο νόημα η Ευρώπη, τότε πρέπει να προωθήσει τις αξίες της. Η Ευρώπη ε, δεν δημιουργήθηκε ως, ως ενιαία αγορά. Ήταν απλώς το μέσο για να δημιουργηθούν ευρωπαϊκές αξίες. Και η συζήτηση για τις αξίες δεν είναι ποτέ ε, εύκολη. Ούτε και στα εθνικά, σε εθνικό επίπεδο είναι εύκολο. Όταν μιλάμε για την ελευθερία της ε, θρησκείας, ε, για την ιδιωτική σφαίρα, οι ίδια δικαιώματα, δικαιώματα γυναικών, δικαιώματα μειονοτήτων, δικαιώματα για τους ομοφιλόφιλους, όλα αυτά είναι δύσκολα και ευαίσθητα και λεπτά θέματα και οδηγούν σε πολύ έντονες ανταλλαγές απόψεων. Αυτές οι εθνικές συζητήσεις τελικά μας οδήγησαν στο να έχουμε κοινέ αξίε στι δικέ μα χώρε. Και αν θέλουμε να προχωρήσουμε την Ευρώπη ακόμα παραπέρα τον 21ο αιώνα, θα πρέπει να έχουμε και κοινέ ευρωπαϊκέ αξίε. Ε, θέλω να μιλήσω σχηματικά. Ε, ε, για μισό αιώνα η Ευρώπη ε, λειτουργήσε με διπλωματικέ διαπραγματεύσει. Πολύ ωραία όλα αυτά. Όσα μιλάμε για ποσοστώσει, για, για γεωργική πολιτική, για διαφορετικά ταμεία, για προπολογισμό. Εύκολα είναι αυτά τα πράγματα. Μπορεί να διαπραγματευτεί κανεί με του εθνικού εκπροσώπου. Ε, μπορεί να γίνουν παζάρια και να δούμε τι εθνικά συμφέροντα ε, διακυβεύονται. Αλλά δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε τις αξίες μας. Δεν μπορούμε να δώσουμε σε μια χώρα ποσόστοση ε, να, ναι, να αντιμετωπίζει με διακρίσει, ας πούμε του ομοφυλόφιλου ή να περιορίζει την ελευθερία του τύπου. Επομένω, οι συζητήσει για αυτά τα θέματα δεν είναι εύκολε, αλλά θα πρέπει να τι κάνουμε αυτέ τι συζητήσει αν θέλουμε να χτίσουμε μια Ευρώπη που μιλάει με μια φωνή προ τα έξω. Αν θέλουμε να έχουμε ε, μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, ειδικά στον τομέα μα, στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Δεν μπορεί να έχεις, φερειπίν πολιτικέ αντιτρομοκρατία χωρί να αντιμετωπίσει το θέμα των αξιών. Δεν μπορεί να έχει ε, ε, συνεργασία δικαστική και αστυνομική χωρί να μιλήσει για αξίε. Ένα απλό παράδειγμα. Στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κάναμε συζητήσει όταν ετοιμάζαμε την απόφαση πλαίσιο για το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Όλοι συμφώνησαν επί της αρχής. Όλοι είπαν είμαστε κατά του ρατσισμού. Όταν μιλάμε για γενικές αρχές, εντάξει όλοι συμφωνήμαστε. Αλλά όταν θέλουμε να τις εφαρμόσουμε αυτές τις γενικές αξίες, ε, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στη συζήτηση για το ρατσισμό και την ξενοφοβία, ένα θέμα αποδείχτηκε πολύ λεπτό. Η άρνηση του ολοκαυτώματος. Σε ορισμένες χώρες είναι ποινικό αδίκημα. Και όμω σε ορισμένες άλλες χώρες το να το καταστήσουμε αυτό παράνομο, την άρνηση δηλαδή, είναι σαν να περιορίσει την ελευθερία του άλλου. Επομένω θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτέ τι αξίε τελικά. Υπάρχουν ε, και πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει, ε, πολύ συγκεκριμένα θέματα στην ατζέντα μα. Ε, σημερινά κράτη-μέλη που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κάποιοι λένε, Κοιτάξτε, η Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση με τι αξίε, με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι εθνικά θέματα αυτά. Εγώ του λέω όχι, δεν είναι αλήθεια. Καταρχά, στι συνθήκε μα ε, έχουμε θεσπίσει τι θεμελιώδει αρχέ και, ελευθε... και αρχέ ε, στο άρθρο 6, όπου βασιζόμαστε. Και για να εξασφαλίσουμε ότι είναι κάτι παραπάνω από ευχολόγια, έχουμε δημιουργήσει και το άρθρο 7 το οποίο είναι το νομικό μέσο και εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να σεβαστούν το άρθρο 6. Και για όσου ε, από εσά δεν είναι ακόμα πεπισμένοι μετά από αυτά που σα είπα, αν πούμε ότι τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα είναι εθνικό θέμα, τότε γιατί ζητάμε από τι υποψήφιε χώρε να σεβαστούν αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γιατί επιμένουμε ότι οι υποψήφιε χώρε θα πρέπει να σέβονται την ε, ελευθερία του τύπου και την ελευθερία του λόγου και δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιβάλλουμε τα ίδια πρότυπα στα σημερινά κράτη-μέλη. Εάν θέλουμε να κρατήσουμε το ηθικό μας κύρος παγκόσμια, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη σέβονται αυτές τις αρχές. Ελπίζω ένας τουλάχιστον να διαφωνήσει με αυτά που σας είπα και ούτω το να για μια συζήτηση, γιατί αλλιώ τι νόημα έχει. Αυτή ήταν η εισαγωγή μου. Κύριε Ισηγητά, χάσατε την αρχή είπαμε να δώσουμε το λόγο για συζήτηση και εσείς ως εισηγητής στο τέλος να κλείσετε αυτή τη συζήτηση και να συνοψίσετε τα όσα διεμήφθησαν. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Έχουμε τον κύριο Ρίτσαρντ Κάλις, ο οποίος ζητάει το λόγο. Πού είστε παρακαλώ, κύριε Κάλιτς. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ σωστά επισημάνατε κι εσείς ότι θα πρέπει να εργαστούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Θα, συμφωνώ, θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σας ότι δεν πρέπει να γίνει συζήτηση. Θα πρέπει ωστόσο να σας πω ότι το όνομα μου Κάλης σημαίνει είναι το όνομα μιας πολιτείας. Ε, υπάρχει μια πολιτεία στην ε, Πολυνία που ονομάζεται Κάλις. 100.000 ε, κατοίκους και άνω έχει. Από την Πολωνία λοιπόν προέρχομαι. Εδώ έχουμε δύο όμω μια πρόταση 24 κρατών που έχουν υιοθετήσει τον χάρτη, τη χάρτα μάλλον των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Από ό,τι φαίνεται η Πολωνία είναι μία από τι τρει χώρε που δεν τον έχει εγκρίνει. Εγώ λοιπόν και η πολιτική μου ομάδα, η αριστερά Συμμαχία της Πολωνίας, διαμαρτυρηθήκαμε για το γεγονός αυτό. Όταν όμως έγινε η διαπραγμάτευση και η προσπογραφή της συνθήκης της Λισαβόνος, η δεξιά είχε την εξουσία στην πατρίδα μου με διάφορες κυβερνήσεις, την ε, πλατφόρμα των πολιτών τώρα, την ε, δικαιοσύνη για τους πολίτες παλαιότερα και διατήρησε αυτή η δεξιά εξουσία την ίδια στάση σε σχέση με το χάρτα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων. Αν μάλιστα πρέπει να έρθει και η συζήτηση στα ανθρώπινα δικαιώματα που η χάρτα χαρακτηρίζει ως θεμελιώδη δικαιώματα. Η Πολωνία, η Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι τρεις χώρες που δεν έχουν υπογράψει αυτή τη χάρτα. Άρα οι πολίτες τους υπολείπονται ω προ την προστασία των δικαιωμάτων του. Δεν είναι ίσοι, δεν είναι ισότιμοι με του πολίτε των λοιπόν κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ίσω όταν έρθει η ώρα να προσφύγουν σε δικαστήρια άλλων κρατών μελών για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά του, θα δούνε τα αποτελέσματα αυτή τη ανισότητα. Συμβολικά, το γεγονό ότι αυτέ οι χώρε δεν έχουν υιοθετήσει τη χάρτα, έχει πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικό το γεγονό ότι δεν έχουν υιοθετήσει τη χάρτα. Όταν λοιπόν μιλούμε για Ευρώπη των πολιτών, όπω ορίζει και ο τίτλο άλλωστε τη σκέψη μα σήμερα, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα ώστε να εξασφαλίσουμε ισότιμα δικαιώματα και ελευθερίε για όλου του πολίτε, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών των, τριών, των τριών κρατών, δηλαδή και τη δική μου πατρίδα τη Πολωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πλατφόρμα, ένα επίπεδο, αν θέλετε, όπου το κάθε κράτο και ο κάθε πολίτης κράτους ή κάτοικος κράτους καλύτερα θα πρέπει να είναι σε θέση να επηρεάζει τις ε, κυβερνήσεις έτσι ώστε να διαφυλάτουν τις ε, πολιτικές ελευθερίες τις ελευθερίες των πολιτών. Στην ε, πατρίδα μου δυστυχώς οι κρατικοί θεσμοί η κρατική εξουσία έχει μεγαλύτερη αξία από ότι ο πολίτης και ιδιαίτερα όταν ε, έχουμε να κάνουμε με την ε, ε, υπηρεσία πληροφοριών, τότε κάθε έννοια προσωπικού βίου και προστασίας του απορρίτου έχει ανατραπεί. Ξέρουμε ότι είχαμε παραδείγματι παράνομες υποκλοπές ακόμη τηλεφώνων δικηγόρων στη χώρα μου. Ε, δεν υπάρχει μάλιστα καμία αιτιολόγηση ε, όπως Φερρυπίν προβολή λόγων κατά καταπολέμησης τρομοκρατίας που θα μπορούσε να αιτιολογήσει ένα τέτοιο Ευχαριστώ λοιπόν πολύ τον, ε, για την έκθεση και νομίζω θα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ε, όταν λέμε... Όταν λέμε... Ευχαριστώ πολύ. Ασφαλώς θα πρέπει να ενταχθεί το θέμα αυτό στην προοπτική της Πολωνίας έτσι ώστε και να υπογράψει τη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κοιτάω το ρολόι, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι δουλεύει όπως πρέπει, αριστερόστροφα δηλαδή. Ίσως έχει πάρει δική του πορεία το ρολόι. Θέλετε εσείς κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ. Η κυρία Μεμετζάν. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω ε, στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στην ε, ε, πρώτη παράγραφο και το, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Η Ευρώπη είναι μια κοινωνία ε, πολλών διαφορετικών πληθυσμών και πολιτισμών ή παραδόσεων. Θα πρέπει λοιπόν να είναι υπερήφανη για την πολιτιστική της ε, πολυμορφία. Ενότητα στην πολυμορφία θα πρέπει να είναι το σύνθημα που θα πρέπει να προβληθεί ακόμη περισσότερο και η έννοια αυτή να χαρακτηριστεί ως θετική διάσταση της Ευρώπης. Την ώρα που αναζητούμε λύσεις θα πρέπει να προβάλλουμε ότι είναι κέρδος η πολυμορφία για μας. Εμείς λοιπόν και ως μέλος της, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης βλέπουμε χαρά ότι δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της αφρομετανάστευσης μέσα στο πρόγραμμα της Στακχόλπ. Θέλαμε για άλλη μια φορά να υπενθυμίσουμε την, την ύπαρξη της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της ε, λαθρομετανάστευσης ε, και το σχετικό σώμα που είναι το μόνο ε, αρμόδιο, το κρέτα το λεγόμενο, ε, να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, με το συντονιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και καλούμε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν, να κυρώσουν τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση σεξουαλικής κατάχρησης και εκμετάλλευση των παιδιών. Και μια και ζητήσατε να συστήσουμε τα θέματα των αξιών και όχι μόνο τα τεχνικά ζητήματα ως εκπρόσωπος υποψηφίου κράτους μέλους, της Τουρκίας δηλαδή, θα ήθελα να πω ότι αυτές οι βασικές ανθρώπινες αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή τα ατομικά δικαιώματα, η δημοκρατία, το κράτος του δικαίου, είναι αυτά ακριβώς που μας ε, προσελκύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας κάνουν να θέλουμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι παράγοντες και σταθερότητα και ασφάλειας και ευημερία για τους πολίτες και εμείς θα θέλαμε να έχουν και οι δικοί μας πολίτες αυτές τις αξίες. Αυτά είναι αξίες σημαντικές και για τους Ευρωπαίους, αλλά και για τους Τούρκους. Πολύ ωραία μας τα είπατε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μορκέτο από την Ιταλία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω πριν από οτιδήποτε άλλο τον κύριο Αγουιλάρ τον οποίο είχαμε συναντήσει και πριν μερικές μέρες στη Γερουσία, στη Ρώμη. Ενθυμούμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση την οποία είχε κάνει. Και εμείς οι γερουσιαστές της Ιταλικής Δημοκρατίας παρακολουθήσαμε με πάρα πολύ προσοχή. Κάποιοι από αυτούς είμαστε σήμερα εδώ, ακριβώς και λόγω της εξαιρετικής ομιλίας του Αγουιλάρ. Πράγματι η ομάδα εργασίας αυτή θα πρέπει να ασχοληθεί με τα ιδανικά και τις αξίες κάτι το οποίο θα ήταν βέβαια πάρα πολύ δύσκολο για όλους όσους συμμετέχουμε. Όταν μιλάμε για ιδανικά και για αξίες, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τις έννοιες αυτές, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανοιχνεύσουμε με ποιο τρόπο εμφανίζονται στο πεδίο της πολιτικής κοινή αυτές οι αξίες και έτσι να καταλήξουμε στη σύμφυση η οποία θα μας επέτρεπε να τις υπακούσουμε αν θέλετε και να τις σεβαστούμε. Κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια σε επίπεδο συναισθήματος όλοι συμφωνούμε. Όταν όμως κυριαρχούν κάποιες λογικές ορθολογικού σε εισαγωγικά τύπου όπου επικρατούν κάποιες κομματικές λογικές, όπου επικρατούν κάποιες διαφορετικές πολιτικές μη πιστοποιημένες από όλους παραδόσεις και συμμερίζομαι εδώ και αυτές τις λεγόμενες χριστιανικές αξίες, τότε η προσπάθεια αυτής εδώ της ομάδας γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε όχι τόσο με ιδέες και με έννοιες, αλλά με συγκεκριμένα πράγματα να φύγουμε από το αφηρημένο και να περάσουμε στο συγκεκριμένο. Έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα μακρόν τα θέματα της μετανάστευσης. Υπάρχουν όμως καταστάσεις όπως στη δική μου χώρα οι οποίες είναι ιδιαίτερα μυστήριες. Εμείς καταλήξαμε σε μια συμφωνία με τη Λιβύη σαν παράδειγμα. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή τα σκάφη μας μαζί με τα σκάφη του Λιβικού Ναυτικού έχουν την δυνατότητα να επαναπροωθήσουν τις φουσκωτές βάρκες οι οποίες προέρχονται από τη Λιβύη και να τις πιέζουμε να επιστρέψουν στη Λιβύη. Αυτό εντάσσεται στα πλαίσια προστασίας των των υδάτων των εθνικών της χώρας μου είναι ένα δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Όταν κάποιος φτάνει παράνομα στα σύνορά του πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τον απομακρύνει, να τον αποτρέψει να εισέλθει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας. Από τη μία λοιπόν πλευρά εμείς πρέπει να εγγυηθούμε το δικαίωμά μας να αποτρέψουμε αυτές τις παράνομες εισόδους, από την άλλη όμως πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να ζητήσουν πολιτικό άσυλο. Πώς θα γίνει αυτό. Εμείς είμαστε επίσης υποχρεωμένοι με τα σκάφη μας να βοηθήσουν, να συνδράμουν αυτούς τους απελπισμένους όταν έρχονται με τα σκάφη τους. Και θα πρέπει να τους ελέγξουμε ταυτόχρονα αν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση χορήγησης ασύλου. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε κάποια κέντρα εντοπισμού, αν θέλετε, των παράνομων αυτών μεταναστών στην ίδια τη Λιβύη. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ξέρουμε ότι αυτοί οι παράνομοι μετανάστες δεν θα παρουσιαστούν σε αυτά τα κέντρα και θα προσπαθήσουν πάλι μέσα από τα πρόχειρα αυτά σκάφη τους παράνομα να έλθουν στη χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία απαιτούν θα έλεγα μια ευρωπαϊκή επεξεργασία από πλευρά της Ευρώπης πολλές φορές μας κατηγορείτε στην Ιταλία. Μας λέτε ότι δεν συμπεριφερόμεθα σωστά απέναντι στους παράνομους μετανάστες. Thank you for that, um, contribution. Mr. Ο κύριος Μπάρκολτ από τη Σουηδία. Unga människor. Och jag tycker det är väldigt viktigt. Πρόεδρε, ευχαριστώ και θέλω να φερθώ περισσότερο στην Ευρώπη των νέων. Οι νέοι πολίτες είναι εκείνοι στους οποίους θέλουμε να παραδώσουμε την κοινωνία μας. Εμείς έχουμε πολύ ε, μεγάλη έμφαση δώσει στους νέους στη Σουηδία και όχι μόνο σε επίπεδο θεσμών. Θέλουμε πιο πολύ να δούνε τι ιδιαίτερα μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. θα πρέπει να ε, τους δείξουμε ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση ασφαλή στο ίντερνετ, θα πρέπει να τους δείξουμε ότι μπορούν να ε, εξασφαλίσουν την προστασία του προσωπικού τους βίου ακόμα και όταν κάνουν ε, περιήγηση μέσα στο διαδίκτυο. Προστασία λοιπόν του ιδιωτικού βίου. Επίσης θα πρέπει να δούμε θέματα αμφιλεγόμενα όπως σε παραδείγματι ε, ζητήματα που έχουν να κάνουν ε, με την αντιμετώπιση αυτής της μορφής ομοιρίας που έχουμε στη σύγχρονη εποχή, δηλαδή τη μάστιγα του ε, εμπορίου ανθρώπων. Έχουμε πολλά φαινόμενα αλληλένδετα μεταξύ τους, γιατί όταν υπάρχει η δυνατότητα αγοράς ή αγοραπολισίας σε ε, υπηρεσίες σεξουαλικού τύπου δεν είναι δυνατόν να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο ανθρώπων. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να αγοράσει κανεί αυτή την υπηρεσία, πάντοτε θα παραμένουν και τα προβλήματα ω προ την ε, εκμετάλλευση των ανθρώπων. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. Χρειάζεται λοιπόν μια νέα στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα βελτιώσουμε την, ε, ε, τι συνθήκε που ισχύουν ως προς την προστασία των παιδιών και ιδιαίτερα και την προστασία των παιδιών από την βία. Και σκοπεύουμε στην ε, Σουηδία να ενισχύσουμε την ε, απαγόρευση μέσα από την νομοθεσία μας της άσκησης σωματικής βίας εις βάρος των παιδιών. Θα ήθελα να εκφράσω εν προκειμένου την ε, ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξη που μας έχει προσφερθεί στην προσπάθεια αυτή. Ξέρουμε ότι πολλά είναι τα κράτη τα οποία ακολουθούν το δρόμο αυτό, της απαγόρευσης δηλαδή της χρήσης σωματικής βίας στις βάρος των παιδιών και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ανοιχτά. Ευχαριστώ. Eh, Σα ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Συμπρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω τόσο είπε η συνάδελφο, ότι έχουμε να κάνουμε την καταπολέμηση του εμπορίου ει βαρό ανθρώπων, τη ε, καταναγκαστική πορνεία και πολλών άλλων προβλημάτων. Εμεί έχουμε στην ε, Σουηδία απαγορεύσει με ποινική κύρωση ε, την αγορά, αγοραπολισία υπηρεσιών γενετήσου χαρακτήρα και θα θέλαμε να μας ακολουθήσουν και άλλες χώρες στην εισαγωγή μιας τέτοιας νομοθεσίας. Νομίζουμε ότι έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα εκμετάλλευση ανθρώπων. Πολλά από τα προβλήματα αυτά δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε μόνο, δεν μπορούμε μόνο να τα προλάβουμε. Θα πρέπει να επιβάλλουμε και ουσιαστικές και ισχυρές κυρώσεις. Για δε τη διεθνή εγκληματικότητα, ήθελα να πω ότι όντω έχουμε κατά προτεραιότητα καθήκον και εμείς ιδιαίτερα οι Σουηδοί της αριστεράς ε, στο ε, Κοινοβούλιο θέλουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη ουσία στα μέτρα τα οποία εισάγονται. Μέσα στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, ωστόσο, δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση για τα μέτρα. Και θα θέλαμε να εξετάσουμε τις ε, επιπτώσεις που έχουν ε, τα μέτρα ή τον αντίκτυπο που μπορεί να, έχουμε, να έχουν κάποια μέτρα. Γι' αυτό θα θέλαμε πριν να προτείνονται νέες λύσεις να εξετάζεται η αποτελεσματικότητά τους. Δεν μπορούμε πάντα να ξεκινούμε με βάση μηδενική. Πρέπει να έχουμε μια βάση από την οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και επίση θα θέλαμε να ορίσουμε και κάποιου όρους, κάποιες συνθήκες προστασίας των θυμάτων της εκμετάλλευσης, ακόμη και πέραν των συνόρων. Άνθρωποι που πέφτουν θύματα εκμετάλλευση είτε σε επίπεδο εθνικό είτε σε επίπεδο ευρωπαϊκό πρέπει να προστατεύονται, είναι τα θύματα. Και η έννοια αυτή τη προστασία αποτελεί για μα ουσιοδέστατο όρο. Αν μου επιτρέπετε, θα αναφερθώ ακόμη σε ένα σημείο τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία έχω τοποθετηθεί και προηγουμένως. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ουσιαστική προσπάθεια για αποτροπή των παραβιώσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε να προστατεύουμε, να προστατεύσουμε τον ιονδήποτε πολίτη από την αρνητική διάκριση που θα του επιβληθεί ενδεχομένως α, λόγω της εθνοτικής του προέλευσης ή λόγω του φίλου του. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, θα επανέλθω στο ερώτημα το οποίο έθεσα στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Έχει ενδιαφέρον να προσπαθήσει να δεις να ξεχωρίσει τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί από τους ομιλητές μέχρι τώρα. Πώς θα αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποια θα είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε σε μια πρώτη φάση για τα θέματα τα οποία έχουμε θέσει. Είναι θέματα τα οποία παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες και σίγουρα θα πρέπει στα θέματα αυτά όχι μόνο να συζητήσουμε αλλά να καταλήξουμε σε κάποιες κοινέ πολιτικές θέσεις. Κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Από την άλλη όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη μια διαδρομή στην προσπάθεια επίλυσης. Ο κύριος Ιωάννης Φίμπνερ από το ε, από την Αυστριακή ε, Βουλή. ανοβούλη Θα ήθελα να αφαιρθώ στις αξίες, ε, κυρία Νοτφέλτ, και τη συζήτηση περί αξιών που βλέπω ότι δεν γίνεται διεξοδικά ως προς τις παραδώσει τα δικαιώματα και τις αξίες. Μιλάτε για τις παραδοσιακές αξίες και την προστασία του πολίτη στην Ευρώπη, την υποχρέωση δηλαδή για το κράτος να διαφυλάξει τη σφαίρα ελευθεριών του πολίτη. Όμως έχουμε κάνει ένα βήμα παραπάνω, όπως, μίλησε και η σας, όπως είπε και η προλαλή σα από τη Σουηδία. Τώρα έχουμε να κάνουμε με τις συσταλτικές αξίες, εκείνες που συστέλουν τις, ε, τα δικαιώματα. Δηλαδή, αναμφίβολα θα πρέπει μια σφαίρα αξιών να παραμένει ουδέτερη ως προς τις αξίες ένα σύνολο αξιών. Όμως όταν πρέπει να επιβληθούν αξίες ε, με την ε, χρήση απαγορεύσεων, τότε περνούμε σε ένα πεδίο αντιπαράθεση, όπως έχουμε δει να συμβαίνει σήμερα. Η περιστολή και μάλιστα με ποινικέ κυρώσεις του ρατσισμού, της ε, ξενοφοβίας, της ομοφοβίας, ε, των σεξουαλικών στερεοτύπων, της προσφοράς ή εξαγοράς ε, γενετήσεων υπηρεσιών, είναι πεδίο περισταλτικών αξιών. Δηλαδή, περιορίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τη μορφή με την οποία ήταν μέχρι τώρα γνωστά. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της διαφύλαξης και επέκτασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και από την άλλη της περιστολής αυτών. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε τον όρο ανάπτυξη ή διεύρυνση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπω γίνεται εδώ στο πρόγραμμα τη Στοκχόλμη. Και γι' αυτό νομίζω ότι η συζήτηση περί αξιών και η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια θα πρέπει να ε, θέσει ένα όριο όπου θα πει μέχρι τώρα αφήναμε τις αυτοεξαγγελθήσεις κοινότητες, δηλαδή κράτη, να προσδιορίζουν το σύνολο αξιών και τα ανθρώπινα δικαιώματα που εφαρμόζουν, ενώ εμείς τώρα έχουμε ξεπεράσει το επίπεδο αυτό και έχουμε φτάσει στο επίπεδο όπου Συμβούλιο και οι λοιποί ορίζουν για τους υπόλοιπους, για το δεύτερο επίπεδο, το τι ισχύει ως ανθρώπινα δικαιώματα. Και επίσης αυτός ο μανδύας της θρησκευτική πίστεως, επί ε, ε, που θέλουν ορισμένοι να χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν ολόκληρο το πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν μπορεί να συνάδει με την ανάπτυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά μόνο με την περιστολή τους. Εγώ προσωπικώς δηλώνω εχθρός της περιστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιστεύω ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη έχουμε μπει σε έναν πολύ οδυνηρό και ακαθόδη δρόμο και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ελένη Φλότρου, παρακαλώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Θέλω να πλειοδοτήσω σε σχέση με αυτά που είπε ο προηγούμενο ομιλητή, σε ό,τι αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών. Γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση στην Ευρώπη για τα δικαιώματα και τι αξίε. Ε, είναι ενδιαφέρον ότι εστιάζεται περισσότερο στις αξίες ε, και λιγότερο στα δικαιώματα. Γιατί τα δικαιώματα ε, μας δεσμεύουν. Μας δεσμεύουν οι συμβάσεις που έχουμε επικυρώσει και αυτό μας ενοχλεί κάπως, ενοχλεί τον κόσμο που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά καμία θεμελιώδης ελευθερία δεν είναι απόλυτη. Η ελευθερία έκφρασης, ε, η ελευθερία η θρησκευτική συνείδηση και σκέψης είναι ελευθερίες οι οποίε ε, δεν είναι απόλυτε, γιατί υπάρχει μια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά τι πρέπει να πούμε, πρέπει να πούμε ότι οι ενδεχόμενε. Ε, οι ενδεχόμενοι περιορισμοί ε, αφορούν κάποιους κανόνες που και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αύριο, μεθαύριο μέσα από τις δεσμεύσεις ε, ε της Χάρτας ε, την 1η Δεκεμβρίου ή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης λαμβάνουν σάρκα και οστά. Αυτό που θα πρέπει να χτίσουμε από κοινού είναι κάποιοι μηχανισμοί που μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε ανεξάρτητα και αντικειμενικά της ε, ελλείψεις και τη μη τήρηση των δεσμευσεών μας, της ε, ελλείψεις μας και πώς θα μπορέσουμε να τις διορθώσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Είπα προηγουμένως ότι δεν είναι δύσκολο το να κάνουμε την τεκμήριωση και νομίζω ότι η η υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, κάνει καλή δουλειά. Θα πρέπει να την ενθαρρύνουμε. Και σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία θα πρέπει να τη δώσουμε ένα πεδίο εφαρμογή, ένα κύκλο αρμοδιοτήτων πιο ευρύ. Και οι συστάσει αυτή τη ε, υπηρεσία θα πρέπει να είναι ε, δεσμευτικέ και να συζητούνται στο Συμβούλιο, στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποχρεωτικά. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε πραγματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο μηχανισμών μας, ως προς το πώς θα εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το τελευταίο σημείο που θέλω να πω. Νομίζω ότι η προσέγγιση για το άσυλο και τη μετανάστευση στο πρόγραμμα της Στοχόλμης δεν είναι η βέλτιστη δυνατή εκ των προτέρων νομίζω ότι δεν έχει νομιμότητα. Η προσέγγιση που θα έπρεπε να έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση είναι αυτή που υπάρχει σήμερα στα πλαίσια του ΟΗΕ που διεκδικούν το δικαίωμα στην κινητικότητα ως το πιο αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμηση της στόχια στον πλανήτη και καταπολέμηση τον φαύλο κύκλο που υπάρχει σε ορισμένες χώρες. Κλιματικά δικαιώματα, ε, έλλειμμα ανάπτυξης, είναι ένας φαύλος κύκλος. Και το ξέρουμε αυτό ότι υπάρχει. Είμαστε τρεις εβδομάδες πριν από την Κοπενχάγη. Ε, Ξέρουμε ότι οι, κλιματικοί κανονισμοί ε, επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους και προκαλούν θανάτους. Μας τα λένε τα Ηνωμένα Έθνη αυτό. Ε, τα Ηνωμένα Έθνη μιλούν για το δικαίωμα της κινητικότητας. Αυτή είναι μια καλή προοπτική. Γιατί, τελειώνω έτσι, γιατί οι μετανάστες που είναι εδώ στην Ευρώπη ε, συνεισφέρουν με θαυμάσιο τρόπο στην ανάπτυξη της χώρας προέλευσης. Πολύ περισσότερο από τις δικές μας πολιτικές ανάπτυξης ε, οι οποίες, ε, μέσα από τις οποίες παζαρεύουμε ένα ή δύο ευρώ παραπάνω. Και δεύτερο, γιατί αυτό το δικαίωμα στην ε, κινητικότητα είναι η απάντηση στη φτώχεια. Αντί να βάζουμε εμπόδια, θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτό το κλάδο της μετανάστευσης. Αυτό όμως δεν, είναι, δεν υπάρχει στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Ε, με αυτό το πρόγραμμα ε, απλώς έχουμε περισσότερη καταστολή και περισσότερη ποινικοποίηση. Ε, κυρία Ιντβέλτ, ε, δεν ήμουν πολύ αυστήρη ε, μέχρι στιγμής. Ε, το ρολόι λέει τα δικά του. Εγώ όμως θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σεβαστείτε το χρόνο που σας έχω δώσει, τρία λεπτά, για να σεβαστείτε και το χρόνο των συναδέλφων σας. Η κυρία Σκέβη Κουκούμα από την Κύπρο είναι η επόμενη μιλήτρια. καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που η Τουρκία αναγνωρίζει την αναγκαιότητα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναμένουμε να περιλάβει και την Κύπρο όταν θα αρχίσει να τα υλοποιεί. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων εγκαθιδρύεται επιτροπή με αποκλειστικό ρόλο των συντονισμών και εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας η οποία όμως δεν θα υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο ενώ επιπρόσθετα αποκλείεται ο δικαστικό έλεγχο των πράξεων που θα λαμβάνουν στον τομέα τη δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων. ο απαράβατο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συνεχής διεύρυνση των πολιτικών ελευθεριών πρέπει δεσμευτικά να είναι ο κοινό παρονομαστή για κάθε κοινοτική και εθνική πολιτική. από την άλλη το φαινόμενο τη μετανάστευση δεν μπορεί να μπαίνει κάτω από το φακό των επιχειρηματικών αναγκών ή να αντιμετωπίζονται οι μετανάστε ω εισβολή στην ευρώπη φρούριων όπω κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν. τα μέτρα καταστολή έναντι των μεταναστών που βλέπουμε να εισάγονται σε πολιτικέ τη ευρωπαϊκή ένωση όχι μόνο καταπατούν διεθνώ κεκτημένα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά αποδεικνύονται και αναποτελεσματικά. η απάντηση στο φαινόμενο αυτό είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτίων τη μετανάστευση η πόλεμη και η φτώχεια δηλαδή σε συνδυασμό με μια ανθρωποκεντρική κοινή μεταναστευτική πολιτική αντάξια των δημοκρατικών παραδόσεων και αξιών των λαών τη υπήρου μα οι εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων οφείλουν να είναι υπερασπιστέ των δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατακτήθηκαν μέσα από σκληρού αγώνε των λαών μα κατά τον περασμένο αιώνα. είναι σημαντικό όμω να υπενθυμίζουμε ότι η ελευθερία η ασφάλεια και η δικαιοσύνη δεν μπορούν να αντικριστούν έξω από την κοινωνικο οικονομική πραγματικότητα. οι ταξικέ ανισότητε η ανεργία οι διακρίσει και η φτώχεια που γεννά το μοντέλο ανάπτυξη τη ευρωπαϊκή ένωση και που θα ενταθεί με τη συνθήκη τη λισαβόνα καθώ και τη στρατηγική αποψηλώνουν τα κατοχυρωμένα δικαιώματα και το επίπεδο ζωής των λαών. γι' αυτό προς τη σημερινή χρήσιμη συνάντηση θα ήθελα να τονίσω ότι για τα προβλήματα και τις ανάγκες των λαών και των εργαζομένων της οπήρους μας οι λύσεις βρίσκονται σε ένα διαφορετικό δρόμο οικονομικής ανάπτυξης που θα βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο του. ευχαριστώ. Όπως είπαμε έχουμε δικαιώματα, έχουμε και καθήκοντα. Έχετε δικαίωμα να μιλήσετε, έχετε καθήκον να τελειώσετε σε τρία λεπτά. Η κυρία Καμί Ιντιού από το Βέλγιο έχει το λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι. Υπάρχουν τρεις βασικές αρχές τις οποίες θα ήθελα να εδράζεται η Ευρώπη. Η ελευθερία, η ισότητα και η αδελφοσύνη. Η ελευθερία έκφρασης δεν έχει νόημα εάν δεν στηρίζεται σε άλλα δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην ιατρική φροντίδα, το δικαίωμα στον πολιτισμό κτλ. Μόνο έτσι μπορεί κανείς να έχει μια αξιόπιστη ζωή σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Αυτό προϋποθέτει την αναζήτηση της ισότητας και ιδιαίτερα εδώ πρέπει να σεβαστούμε το δικαίωμα στην απασχόληση, το δικαίωμα στην εργασία, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα δυστυχώς στο σύνολο της Ευρώπης. Και αυτό είναι κάτι που εμπλέκει αν θέλετε πέραν των πολιτικών και την ευθύνη των εταιριών, των επιχειρήσεων, των ιδιωτικών εταιριών. Ξέρουμε ακριβώς πώς γίνονται κάποιες μετακινήσεις εταιριών στο εσωτερικό της Ευρώπης και εκτός αυτής και ξέρουμε ότι έτσι τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν γίνονται σεβαστά. Και γι' αυτό ακριβώς είχα καταθέσει κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας, για τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας, το δεύτερο εξάμεινο του 10 δηλαδή, μία πρόταση έτσι ώστε να υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα εγγυημένο διεπαγγελματικό εισόδημα. Δεν σας δίνω τεχνικές λεπτομέρειες σε αυτή τη φάση, αλλά υπάρχει δυνατότητα να το επιδιώξουμε και να το πετύχουμε. Να σας θυμίσω αυτό που έλεγα προηγουμένως. Πρέπει να επιδιώξουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεταναστών που έχουν εγκατασταθεί επίσημα στην Ένωση. Νομίζω ότι η πρόσβαση σε αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα θα ρυθμίσει τα πολλά προβλήματα που έχουμε μεταξύ μας, προβλήματα που άπτονται και του οργανωμένου εγκλήματος. Έχω την αίσθηση ότι οι συμπολίτε θα πιστέψουν στην Ευρώπη τη στιγμή που η Ευρώπη θα λάβει τις συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες θα τους βοηθήσουν. Να πω επίσης ότι οι οδηγίες σαν και αυτές που γνωρίσαμε στο παρελθόν, η οδηγία Μπολκενστάιν ή η, η, η οδηγία για την πλήρη απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι ερωτηματικά μεγάλα γιατί η Ευρώπη εδώ πρέπει να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Σας ευχαριστώ. Ήσασταν ιδιαίτερο σύντομοι. Ο Λόρδος Μακλέναν έχει το λόγο. Πρόεδρε. Η εποχή μας ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να αναζητήσουν συνεργασίες διαμεθοριακές, να διευκολύνουν και να δώσουν εγγυήσει για τη σωστή καταπολέμηση του εγκλήματος. Έχουμε ακούσει αρκετά για το θέμα αυτό και στα πλαίσια της καταπολέμησης των ναρκωτικών και της τρομοκρατίας. Δεν ακούμε όμως πάρα πολλά για την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών σχετικά με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του εγκλήματος και στον τομέα της αναλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται ε, με την επιβολή του νόμου και της τάξης. Έχω εντυπωσιαστεί μέχρι τώρα από την έκθεση η οποία κυκλοφόρησε πριν από αυτήν τη συνάντηση και προέρχεται από τον ελεγκτή της προστασίας προσωπικών δεδομένων, τον κοινοτικό ελεγκτή. Συμπερασματικά θα έλεγα στην τελευταία του έκθεση που κυκλοφέρισε τον Ιούλιο και ε, σχολιάζει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη φάση αυτή που συζητάμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και στη φάση αυτή όπου περιμένουμε άμεσα τη συνάντηση κορυφής του Συμβουλίου να υπογραμμίσουμε την μεγάλη σημασία που έχει η βασική αρχή προστασίας των πολιτών προσωπικών δεδομένων, μια βασική αρχή η οποία θα πρέπει να συμπεριληφθεί σαφώς και σε κάθε νομοθετική πρόταση η οποία θα θεωρηθεί σημαντική για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Τον Ιούνιο του 2008 το Συμβούλιο αποφάσισε για μέτρα διαμεσοριακής ε, συνεργασίας σε περιορισμένο όμως επίπεδο. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλά, ιδιαίτερα στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσει κανείς την κριτική την οποία ασκεί ο ελεγκτής προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εντοπίζει τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν για τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου ανταλλαγής πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι και στο μέλλον οι περιοριστικοί όροι θα πρέπει να είναι κατευθυντήριοι όροι θα έλεγα για τα συστήματα λειτουργίας ανταλλαγής πληροφοριών. Κάτι το οποίο και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω σαφώς το έχει στο κέντρο της προβληματικής του ιδιαίτερα από την 1η Δεκεμβρίου μετά την εφαρμογή της συνθήκης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τίσιο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε ε, να μιλήσω. Θα ήθελα να εστιάσω σε ένα πράγμα. Με χαροποιεί το θέμα που θέσαμε σήμερα ε, ως θέμα συζήτησης. Γιατί σε προηγούμενες φάσεις, όταν δουλεύαμε για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, για τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, δεν συζητήσαμε ποτέ τις αξίες. Ε, και δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε όμως ε, ποια είναι η σχέση αξιών και δικαίου. Οι αξίες είναι τα θεμέλια του δικαίου και το δίκαιο ε, δημιουργείται για να προστατευτούν οι αξίες. Επομένως, νομίζω ότι είναι κρίμα που στις δύο νομοθετικές διαδικασίες που ανέφερα δεν υπήρχε καμία αναφορά στο Θεό από την οποία εκπορεύονται κάποιες αξίες και στις χριστιανικές αξίες που να μην ξεχνάμε ότι είναι τα θεμέλια για τους ιδρικούς, ιδρυτικούς πατέρες της Ευρώπης, ε, για τον Γκάσπαρη και για τον Σούμαν. Ε, σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα θεμελιώδες ερώτημα. Ποιες είναι οι αξίες που θέλουμε να προστατεύσουμε. Γιατί οι αξίε αυτές δεν είναι διαχρονικές, δεν είναι υπερβατικές. Τι είναι, είναι το αποτέλεσμα μιας ψήφου, το αποτέλεσμα των ψήφων στην ιστορία μα, μας οδήγησε στην εφαρμογή και πολλών αρνητικών νόμων για τους οποίους αργότερα ντρεπόμασταν. Επομένως, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μια κατάσταση όπου τα διεθνή δικαστήρια ψάχνουν να βρουν λύσεις οι οποίες δεν είναι πολύ ευτυχείς. Ε, γι' αυτό λοιπόν η Πολωνία έχει τις επιφυλάξεις ό,τι αφορά τον δεσμευτικό χαρακτήρα της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, από μόνο το αυτό το κείμενο είναι πολύ όμορφο. Και καλό είναι στην Ευρώπη να έχουμε τόσο υψηλέ και ευγενεί φιλοδοξίε. Αλλά από τι πρόσφατε αποφάσει του Δικαστηρίου του Στρασβούργου βλέπουμε ότι συχνά εφαρμόζεται η τέταρτη γενιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Πολωνία έχει δυσπιστία απέναντι σε τέτοια ε, δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη από τα ομοφιλόφιλα ζευγάρια κτλ. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ε, απειλές που υπάρχουν ε, στην προσπάθεια ανάπτυξης των ε, θεμελίων και αξιών της Ευρώπης. Καλό είναι να στραφούμε λίγο προς το παρελθόν για να εμπνευστούμε για το μέλλον. Ευχαριστώ. Σω το λόγο στον επόμενο μιλητή να τονίσω ότι μία από τις βασικές αξίες της Ευρώπης είναι η ελευθερία της συνείδησης. Όταν δημιουργήσαμε αυτή τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ε, είχαμε στο μυαλό μας την ελευθερία συνείδησης και τη σκεφτική ελευθερία. Εγώ ως φιλελεύθερη και άθεη αυτές τις ελευθερίες ε, προωθώ. Και διαφωνώ κάθετα, αγαπητέ κύριε, ότι η θρησκεία έχει το μονοπόλιο στην ηθική. Νομίζω ότι και οι άθεοι έχουν ε, ηθικές αξίες και ρίσματα. Ελπίζω να το σεβαστείτε αυτό, το δεχτείτε αυτό σε μια ένωση τόσο ποικιλόμορφη. Εγώ σέβομαι τι απόψει σα και τη θρησκεία σα και τη συνείδησή σα. Θα ήθελα και εσεί να σεβαστείτε τη δική μου. Γι' αυτό χαίρομαι που δεν υπάρχει καμία αναφορά στο Θεό, ε, ούτε στο Σύνταγμα, ούτε στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Γιατί αυτό θα απέκλειε πάρα πολλού ανθρώπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο πάντων, τώρα, μετά από αυτά, νομίζω ότι ο κύριο Σένα από την Αυστρία έχει τον λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα τελευταία σας λόγια. Ήταν τα σωστά λόγια την κατάλληλη στιγμή. Και αυτό ακριβώ εδώ είναι και το ενδιαφέρον. Η ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ξεκινάει με την Αμερικανική Επανάσταση και δύο-τρία χρόνια μετά στο Παρίσι με τη Γαλλική Επανάσταση και εμείς οι Ευρωπαίοι την έχουμε αναπτύξει με τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα δικαιώματα της γυναίκας. Εκλέγην και εκλέγεστε για τη γυναίκα. Όλα αυτά γίνανε στην πορεία μιας εξέλιξης. Ο κίνδυνος τώρα είναι να πούμε προστασία των πολιτών μένα, αλλά στην πραγματικότητα, μέσα από μια οργουελιανή πραγματικότητα, να αρχίσουμε από μέσα να περιστέλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν λέμε θέλουμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, πρέπει να αποφύγουμε να εξασφαλίσουμε, να, να επιτρέψουμε τη νίκη για ακριβώς αυτούς τους τρομοκράτες, γιατί αυτό θέλουν οι τρομοκράτες, να μας εξαναγκάσουν να περιορίσουμε τα δικαιώματά μας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα-ένα κομμάτι-κομμάτι, βήμα-βήμα. Αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε και εδώ ακριβώς είναι και το συγκλονιστικό αυτής της πορείας και γι' αυτό και εγώ αγωνίστηκα μέσα από τη διαδικασία της συνθήκης Λισαβόνας ότι έχουμε εδώ κοινέ θεμελιώδεις αξίες, θεμελιώδη δικαιώματα έχουμε μία παράδοση μοναδική όπου το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβάλλει τον σεβασμό των δικαιωμάτων. Έχουμε καταδικάσει την ε, ομοφοβία, το, τη θανατική καταδίκη, την παραβίαση των δικαιωμάτων, την παραβίαση των δικαιωμάτων ή την, ε, τις διακριτικές μεταχειρήσεις εις βάρος ορισμένων πολιτών. Όλα αυτά τα έχουμε εξασφαλίσει. Αλλά τώρα κινδυνεύουμε να πούμε θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, αλλά διαφοροποιώντας μεταξύ εκείνων για τους οποίους δίνεται η δυνατότητα γιατί έχουν την ηθαγένεια και μεταξύ των άλλων που ζουν στις χώρες μας και δουλεύουν στις χώρες αυτές αλλά δεν έχουν τέτοια δικαιώματα και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει ακόμη περισσότερο να επεκτείνουμε την ε, πρόταση της Στοκχόλμης και ιδιαίτερα τη συνθήκη του Δουβλίνου. Διότι είναι αδιανόητο να υπάρχει, μόνο οι οικονομικοί λόγοι μπορεί να εξηγούν μια τέτοια διαφορά, μια τέτοια απόκληση, να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στις χώρες μας και νόμιμα, αλλά δεν έχουν τέτοια δικαιώματα με μας. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε μια τραγωδία όχι μόνο ανθρώπινη. Έχουμε να κάνουμε και με μια τραγωδία οικονομικών διαστάσεων. Οι συνέπειες της ζωής των ανθρώπων αυτών. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ προηγμένη πολιτική γειτονία η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσαμε να μεριμνήσουμε και στον τομέα αυτών και πέραν των όριων του Σέγγεν να ενισχύσουμε και την κοινωνική ενσωμάτωση και το πεδίο της προκοινωνικής προστασίας. Η κυρία Βέρτσμαν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε αρκετά από τα σημεία θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Ιδιαίτερα θα ήθελα να υπογραμμίσω τα δικαιώματα των παιδιών. Στην πατρίδα μου από, τις, το σημερινό τύπο βλέπω ότι μόνο 20 χρόνια μετά τη θέσπιση της δημοκρατίας αναγνωρίστηκαν τα δικαιώματα των παιδιών σε συνταγματική διάταξη. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση προ προστασία των παιδιών και θα ήθελα και όλα τα κράτη να υιοθετήσουν το χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα τη χάρτα των δικαιωμάτων των παιδιών και να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα αυτά απολύτω. Και λόγω και τη επικαιρότητα τη χώρα μου θα ήθελα να επισημάνω ένα ιδιαίτερο σημείο που αφορά την ισότιμη μεταχείριση και τι ισότιμε δυνατότητε για τι γυναίκε. Εγώ δεν μπορώ να χαρακτηριστώ ω φεμινίστρια μαχόμενη, αλλά όταν για την ίδια δουλειά η γυναίκα παίρνει λιγότερο λιγότερα χρήματα. Μερικέ φορέ ο μισθό τη είναι και 25% χαμηλότερο από του αντίστοιχου άντρα συναδέλφου του. Διαρωτώ με τι είδου δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε και τι είδου διαφύλαξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων μα προσφέρει η Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να μεριμνήσουμε, να τα προαγάγουμε και μέσα στην τρέχουσα θητεία. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ προσυπογράφω τα όσα είπατε. Πριν όμω δώσω το λόγο στην κυρία Λόσο, Α, η κυρία Όλσον όμω μίλησε νωρίτερα, έτσι δεν είναι. Θα ήθελα όμω να επισημάνω ένα σημείο για όλου του συναδέλφου. Οι κυβερνήσει μα, οι κυβερνήσει σα, ε, προετοιμάζουν τώρα την υποψηφιότητα για του υψίστους φόκου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή του 27 επιτρόπου, τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον έχουμε ήδη ορίσει, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου έχει οριστεί. Α, ναι, έχουμε και τον εκπρόσωπο, ε, τον τσάρο των εξωτερικών, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση λίγο μιλήτρια. Και μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε μόνο τρει γυναίκε υποψήφιε. 10% είναι αυτό. Τρει μόνο. Και νομίζω ότι είναι αξιοθρύνητη αυτή η κατάσταση. Θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερο, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έρχεται να ψηφίσει ω σύνολο το, ο, ε, το συλλογικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ προσωπικώ δεν είμαι διατεθειμένη να εγκρίνω συλλογικό όργανο το οποίο περιλαμβάνει μόνο τρει γυναίκε υποψηφίου και νομίζω ότι και εσείς θα μπορούσατε να ενισχύσετε πίεση στις κυβερνήσεις σα να προαγάγουν θέσεις τη γυναίκα και σε, αυτούς τους, σε αυτά τα αξιώματα τα ευρωπαϊκά. Η κυρία Όλσον τώρα νομίζω θέλει να λάβει το λόγο για δεύτερη φορά. Πρόεδρε, δεν μπορώ να λάβω το λόγο για δεύτερη φορά. Έχω ήδη μιλήσει. Βέβαια. Ναι, ναι, μπορείτε, λέει η Πρόεδρο, αλλά υπάρχουν και άλλοι που περιμένουν να λάβουν το λόγο. Μια και η δεύτερη σα παρέμβαση, όσο μπορούσατε να είσαστε πάρα πολύ σύντομοι. Ε, Καλώ λέει η κυρία Όλσον, τότε παρετούμε από το δικαίωμα του λόγου. Όχι, όχι, μπορείτε να μιλήσετε, μπορείτε, αλλά να έχετε υπόψη ότι περιμένουν και άλλοι στην ώρα. Καλώς πρόεδρε, εγώ υπόσχομαι ότι δεν θα ζητήσω και τρίτη φορά το λόγο. Λοιπόν, έγινε ο λόγος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άκουσα την κυρία Κουκουμά εδώ, Κουκουμά εδώ από την Κύπρο. Άκουσα την εκπρόσωπο του Βελγίου, οι οποίε εκφράστηκαν με μεγάλη εφράδια και είπαν ότι πρέπει και τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως και τα δικαιώματα των παιδιών ιδιαίτερα, να προστατευθούν. Και θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα, να επανέλθω σύντομα στο θέμα του ασύλου στο κόμμα μου, στο κοινοβούλιο μου, έχει εκφραστεί επανειλημμένως επίκριση, επικρίσεις και μάλιστα εδώ έχω να σας πω ότι έχουμε να κάνουμε μια θέση ιδιαίτερα προηγμένη της γυναίκας στη χώρα μου. Έχουμε όμως προβλήματα όπως η φτώχεια, όπως οι κλιματικές αλλαγές, επιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Και η πολιτική που αναπτύσσεται δεν λαμβάνει υπόψη τη θέση της γυναίκας και του παιδιού. Βλέπουμε, Φερρυπίν, οι επιχειρήσεις επιβάλλουν πολιτικές και το βλέπουμε αυτό και από τις διατάξει του Δουβλίνου οι οποίες έχουν σαν συνέπεια πλέον να είναι αδύνατη η νόμη μεταμονάστευση προς την Ευρώπη. Ή βλέπουμε επίσης ότι η Frontex επιβάλλει πιέσεις βάρος των ανθρώπων, τους πιέζει όλο και περισσότερο να εκτίθενται σε, φυσικό σε σωματικό κίνδυνο προκειμένου να μεταναστεύσουν και πράγμα, αυτό το πράγμα το βρίσκω απόλυτα λυπηρό. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. Και εγώ καλωσορίζω την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει ένα χώρο ελευθερίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πάνω απ' όλα την ασφάλεια των πολιτών μας και τα δικαιώματα των πολιτών μας. Αυτή θα πρέπει να είναι η κύρια μέρημνα, μεριμνά μας. Είμαι η νεαρότερη βουλευτή στο Αυστριακό Κοινοβούλιο και χαιρετίζω τα δικαιώματα των παιδιών, των γυναικών, των νέων που, που αναφέρθηκαν. Ε, όπως είπε και ένας ομιλητής, ε, χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να εγγραφούν στο Σύνταγμα τα δικαιώματα αυτά. Τώρα αυτό το δικό μα Σύνταγμα εννοώ τη Αυστρία. Και αυτό θα πρέπει να συμβεί ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι νέοι έχουν δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Ε, μιλάμε με διάφορα ευχαλόγια. Μιλάμε, λέμε ότι οι νέοι είναι το μέλλον τη Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Να τα κάνουμε αυτά πραγματικότητα. Τώρα, για το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη. Ε, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το πρόγραμμα αυτό. Είναι δύσκολο να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας για τους πολίτες, από τη μία, αλλά μη περιορισμό των δικαιωμάτων τους από την άλλη. Και υπάρχουν διάφορα θέματα που πρέπει να επισύρουν κριτική στο πρόγραμμα της Στοκόλμης, ειδικά σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων. φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν ανταλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, τόσο ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν σωστοί έλεγχοι και σωστή ισορροπία ούτως ώστε οι πολίτες απολάβουν ένα κάποιο επίπεδο προστασίας και ότι τα δικαιώματά τους γίνονται σεβαστά. Δεν θα πρέπει να πέσουν θύματα χρήσεων οι πολίτες μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σεφσικ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα κάνω λίγες παρατηρήσεις σχετικά με αυτά τα οποία άκουσα μέχρι τώρα περισσότερο. Υπάρχει μια τάση, θα έλεγα, ε, συζήτησης και αιμονή σε κάποια θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Στοχόλμης. Εγώ έχω, έχω μιλάμε ας πούμε για το δικαίωμα στην εργασία ε, συζητάμε το θέμα της δικαίωμα, του δικαιώματος στην εργασία ή του καθήκοντος αν θέλετε για εργασία αλλά καλύτερα θα έπρεπε να συζητάμε θέματα ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει λοιπόν να σας προειδοποιήσω ότι αρκεί να μην υπάρχουν διακρίσεις, αρκεί να υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός, αρκεί να υπάρχει δικαίωμα επιλογής και ε, να είναι κανείς αρκετά ανταγωνιστικός για να πάρει τη θέση εργασία την οποία μπορεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Μιας και συζητάμε για αξίες, ε, η βασική αξία για μένα είναι η ελευθερία. Αυτός είναι ο τέος τρίτος πυλώνας, αν θέλετε, του ευρωπαϊκού νομικού, της ευρωπαϊκής νομικής αρχιτεκτονικής. Βασική ελευθερία είναι η ελευθερία επιλογής και για να το κάνει κανείς αυτό πρέπει να είναι κυρίαρχα ανταγωνιστικός και έτσι θα διασφαλίσουμε και μέσα από την εργασία της σταθερότητας της οικονομίας μας θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι ανθρώπινο για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν, για αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη να δουλέψουν και όχι για τους τεμπέληδες. Η αλληλεγγύη δεν είναι ε, κάτι το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αυτούς οι οποίοι λειτουργούν αντικοινωνικά. Ο κ. Αλευράς. Ε, ε, θα ήθελα να πω ότι κατά την άποψή μου η συζήτηση πάνω στις αρχές είναι χρήσιμη και ευχάριστη αλλά εκείνο το οποίο έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανάγκη είναι τα συγκεκριμένα μέτρα. Να συζητήσουμε πάνω σε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας προσώπων που ζουν στις γκρίζες περιοχές του συστήματός μας. Αυτό το οποίο θεωρώ τούτη την ώρα εξαιρετικά κρίσιμο είναι ότι υπάρχουν κατηγορίες του πληθυσμού του ευρωπαϊκού πληθυσμού οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες πραγματικές και κοινωνικές πρόσβασης στα αγαθά του νομικού μας συστήματος ή στις κοινέ αξίες αυτού του συστήματος. Για παράδειγμα, εντός λίγων ημερών στην πατρίδα μου πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη κατηγορούμενου για εκμετάλλευση παιδιών, ξεκινησει η δικη κατηγορουμενων για κακοποίηση δίκη στην οποία κατηγορούμενοι είναι οι γονείς και εκείνοι που κακοποιούσαν. Τα παιδιά στερούνταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της δυνατότητας να αντλήσουν ωφέλη από το νομικό σύστημα. Γιατί υπάρχει στα ευρωπαϊκά νομικά στάνταρτς κάποια πρόβλεψη για αυτές τις κατηγορίες των πολιτών υπάρχει πρόβλεψη για τους πολίτες οι οποίοι ζώντας σε κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να αντιπροσωπευθούν νομικά στο δικαστικό σύστημα, στο δικαιικό σύστημα και να έχουν προστασία. Υπάρχει αξιολόγηση, υπάρχουν δείκτες μέτρησης των νομικών μας συστημάτων οι οποίοι θα επιτρέψουν να σημειώσουμε τις ανεπάρκειες του νομικού μας συστήματος, του δικαιικού μας συστήματος και ταυτόχρονα να τις θεραπεύσουμε. Υπάρχουν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας μηχανισμοί οι οποίοι επιτρέπουν και προσφέρουν προστασία για πολίτες διαφορετικών χωρών οι οποίοι ζουν σε καθεστώς οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Παράδειγμα, μπορώ εγώ πολίτης μιας χώρας ζώντας σε μια άλλη χώρα να έχω ευκολία πρόσβαση στο δικαιωτικό σύστημα όταν δεν έχω τα οικονομικά μέσα δεν γνωρίζω καλά τη γλώσσα και ενδεχομένως ζω υπό καθεστώς οικονομικής εκμετάλλευσης. θεωρώ λοιπόν ότι όσο δεν συζητάμε για τα συγκεκριμένα αυτά μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματός μας όχι στο επίπεδο των αξιών και των αρχών αλλά στο επίπεδο της προστασίας τους εκεί συνεχίζει να υπάρχει ένα Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ. Αυτό ακριβώς του είδους τα θέματα συζητάμε όλο και περισσότερο και με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, νομίζω ότι θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Νομίζω. Τελευταίος ομιλητής, η κυρία Πάρκχολτς. Ευχαριστώ. Μιλάω για δεύτερη φορά και σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Εδώ μιλήσαμε για ένα θέμα αξιών. Εγώ είμαι φιλελεύθερη και φεμινίστρια. Διέκοψε ο πρόεδρος. Μα είναι φυσικό που σας δίνουμε δυο φορές το λόγο, διότι είναι η Σουηδική Προεδρία στη μέση. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ που το θίξατε κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό εν ώψη του μέλλοντος της Ευρώπης. Θα πρέπει να υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και ίση εκπροσώπηση διότι και οι γυναίκες πρέπει να συμμετέχουν στις πολιτικές διεργασίες. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε οι χώρες μέλη να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να συμμετέχουν όχι μόνο διότι θέλουμε στα δημόσια αξιώματα να είναι μισοί άντρες και μισές γυναίκες. Όχι, θέλουμε οι γυναίκες να αποφασίσουν στα σοβαρά. Για το πρόγραμμα τώρα της ε, Στοκχόλμης, βία κατά των γυναικών. Τι μπορούμε να κάνουμε για να παλέψουμε κατά αυτού του φαινομένου είναι ένα θέμα το, οποίο ασχολήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες να μιλήσουμε για το πρόβλημά τους. Οι γυναίκες που υπήρξαν αντικείμενο βίας να ξέρουν ότι δεν είναι μοναχές τους, ότι έχουν μια υποστήριξη για να βγουν από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και τώρα θέλω να, κάνω εδώ, να, εκφέρω μια τρίτη σκέψη. Ορισμένοι ομιλητές είπαν πόσο σημαντικό είναι να ληφθούν ως βάση οι χριστιανικές αρχές. Εγώ όμως βρίσκω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα μεταξύ της ισότητας των γυναικών και των χριστιανικών αρχών και σε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να υπερέχουν η ισότητα ανδρών και γυναικών έναντι της χριστιανικής θρησκείας. Είναι είπα το θέμα, το θέμα της ισότητας και η Ισπανική Προεδρία θα το έχει και στην καρδιά της Προεδρίας της. Σημαντικότατα λοιπόν όλα όσα είπατε και θα τελειώνουμε με τον Αντρέη Γκρζίπ πρόεδρε, πρόεδροι μάλλον. Και αναφέρομαι εδώ στους ε, δύο συμπροέδρους. Ήθελα να πω στη Σουηδική Προεδρία ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ σημαντικό και θα αποτελέσει μια νέα φάση. Πρέπει να έχουμε όμως συνέστηση δύο πραγμάτων. Από τη μια έχουμε πρόοδους στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Απ' την άλλη μεριά όμως το πρόγραμμα αυτό θέτει και περιορισμούς. Άμα πρέπει να εγγυθούμε εμείς την εσωτερική ασφάλεια υπάρχουν στοιχεία εδώ που μας περιορίζουν ως πολίτες. Η απειλή της τρομοκρατίας έχει γίνει, είναι πλέον καθημερινότητα και ταυτόχρονα αυτή η απειλή μας δημιουργεί και ορισμένους περιορισμούς. Το βιομετρικό διαβατήριο είναι θετικό ή είναι ένας περιορισμός των δικαιωμάτων του ατόμου. Για το άτομο σίγουρα είναι περιορισμός γιατί πρέπει να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για μας τους ίδιους. Αλλά για την ασφάλεια σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα διότι εγκιάται την ασφάλεια και όταν μιλάμε για δικαιώματα θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και περιορισμούς. Τώρα για τη μετανάστευση εμείς μιλάμε εδώ για εναρμόνιση του δικαιώματος ασύλου αλλά απ' την άλλη μιλάμε και για ε, μια ασφαλή Ευρώπη. Άμα δεν περιορίσουμε εμείς τη μετανάστευση τότε θα έχουμε και μερικές ε, απρόοπτες συμπεριφορές των γειτόνων μας και κυρίως οι νότιοι ε, τα, μέλη της Ένωσης από τον Νότο ξέρουν πολύ καλά ποια απρόοπτα μπορούν να προκύψουν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια εξυγίανση ε, διότι αυτή η φυσική μετανάστευση η οποία έχει να συνδέεται με τη φτώχεια, με τη λειψιδρία, με τα κλιματικά προβλήματα, με την πείνα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, δρώντας εκεί που το, στις ρίζες του κακού, εκεί όπου υπάρχουν ε, πόλεμοι, καταστροφές κλπ. Οι γείτονες. Εμείς ως Πολωνία ε, γειτνιάζουμε με, τις, με χώρες Σέγγεν και είναι πολύ εύκολο για μας να κυκλοφορούμε αλλά οι γείτονε μας, οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι πιστεύουν ότι ξαναφτιάχτηκε ένα παραπέτασμα. Θέλουμε λοιπόν εμείς να εγγυθούμε αυτές οι χώρες να έχουν μία επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία ανθρώπινη επαφή ε, περάσματος συνόρων αλλά θέλουμε από την άλλη μεριά και ασφάλεια στα πλαίσια του Σέγγεν. Αυτές είναι βασικές αρχές, γιατί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μιλάμε πάρα πολλές φορές για θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν μόνο στο δικό μας εσωτερικό καλό. Αλλά γύρω από τα σύνορά μας δεν υπάρχει το κενό. Υπάρχουν και άλλες χώρες που θέλουν να ζήσουν εξίσου καλά όσο και εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας για να απαντήσει στις παρατηρήσεις που έγιναν. Merci. Gracias. Gracias. Ευχαριστώ όλους και όλα τα μέλη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων που συμμετείχαν στη συζήτηση. Ήταν πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και θα πρέπει να είναι και χρήσιμη. Σε παλιές μας συζητήσεις τα μόνιμα στοιχεία που είχαμε για το θέμα της, του συνδυασμού αλληλεγγύης, ισότητας, αδελφότητας, δικαιοσύνης, πλουραλισμού ε, ως, ε, θεμε... ως ιδρυτικές αξίες μιας ε, ελευ... τάξεως ελευθερίας αναφέρθηκαν πάρα πολλές φορές και αναφερόντουσαν πάρα πολλές φορές συνδεόμενες όμως πάντοτε με τα συντάγματα τα οποία βρισκόταν πίσω από κάθε ε, ε, εθνικό σύστημα. Σήμερα η Ευρώπη δημιουργεί ένα νέο κοινό παρανομαστή χωρίς όμως να καταργεί τίποτα. Τα συντάγματά σας δεν πρόκειται να χαθούν, ε, δεν πρόκειται να, να, διαλυθούν μέσα σε αυτήν την συνταγματική διάσταση, την νέα συνταγματική διάσταση της Ευρώπης. δεν διαλύονται μέσα σε αυτό. Ίσα ίσα το αντίθετο. Πολλαπλασιάζονται, εμπλουτίζονται. Άρα βελτιώνονται και μα ε, και μας βελτιώνει ως πολίτες εμάς τους ίδιους Ισότητα λοιπόν βάσει των κοινών μας συνταγματικών αρχών βάσει της συνταγματικής εμπειρίας της κοινή συνταγματικής εμπειρίας στην Ευρώπη. Και αυτές οι τοποθετήσεις που ακούσαμε σίγουρα μπορεί να υπάρχουν διαφορές αλλά Εκείνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι ότι πέρασαν 10 χρόνια όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση και τη συνταγματική σύγκληση και τελικά αυτές, αυτά τα 10 χρόνια πλέον συγκλίνουν στη συνθήκη της Λισαβόνας η οποία θα αρχίσει να ισχύσει. Πρέπει να κλείνουμε λοιπόν αυτή τη σελίδα και να ορίσουμε αυτόν τον νέο κοινό παρανομαστή δικαιωμάτων και ελευθεριών που είπαμε δεν διαλύονται, δεν χάνονται. όλες οι εγγύησει που έχει κάθε πολίτης όντας πολίτης ενός κράτους μέλους πολλαπλασιάζονται με μια νέα κλίμακα, με ένα νέο επίπεδο προστασίας, με μια νέα ε, κοινότητα δικαίου, με νέες εγγύησει. Αποτέλεσμα αυτών των δέκα ετών συζήτησης για τη Λισαβόνα είναι η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπήρξαν συνταγματικές δυσκολίες στο να την ενσωματώσουμε στη συνθήκη. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αποτελεί μία από τις τρεις συνιστώσεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Έναν ορισμό της συνθήκης, μία χάρτα η ίδια η συνθήκη, το κόρπους της συνθήκης και η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. όπου ορίζεται ένα νομικά δεσμευτικό ηθικό μίνιμουμ της αρχής της ηθαγένειας. και αυτός ο δεσμευτικός ορίζοντας της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί υπόσχεση, βελτίωση αυτού του καθεστώτος του πολίτη στα κράτη-μέλη. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο θα εξελιχθεί θετικά και θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Ακούσαμε στις τοποθετήσεις διάφορες αναφορές σε ετερογενή προβλήματα τα οποία σίγουρα υφίστανται μέσα σε αυτήν την οικοδόμηση του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας, ασφάλειας. Το 1992 με τον τρίτο πυλώνα στο Άμστερνταμ ξεκίνησε. Συνεχίστηκε με το Τάμπερ, εμβαθύνθηκε στη Χάγη και τώρα θα γίνει με τη Στοκχόλμη το ποιοτικό άλμα. Δεν πρόκειται λοιπόν ο χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης και λοιπά να παραμείνει διακυβερνητικός. Αλλά ευρωπαϊκός χώρος όπου θα νομοθετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μόνιμη συνεργασία και διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια. Για ένα σωρό προβλήματα, προκλήσεις κλπ. Διότι τα κράτη-μέλη όλα δημοκρατικά και όλα περήφανα για τη συνταγματική τους ε, παράδοση τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν ότι τους διαφεύγουν όλα αυτά τα προβλήματα, διαφεύγουν από τη δυνατότητα που έχουν να απαντήσουν. Όχι μόνο οι εθνικές